Αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω εγκαρδιότατα στην σημερινή μας συνεδρία της Επιτροπής ΚΡΙΣ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σήμερα καταρχήν μια συνεδρίαση του συνόλου της Επιτροπής μας Παρόλο που κατά βάση εγώ βλέπω μόνο τους ε, συντονιστές και τους εκπροσώπους τους. Λοιπόν, καταρχήν θα έχουμε τις συνεδρίες της Επιτροπής μας που είναι δημόσια. Γι' αυτό χαιρετίζω και όλους τους επισκέπτες που είναι παρόντες. Κατόπιν όμως θα έχουμε και κλεισμένων των θυρών τη συνεδρία των συντονιστών. Πήρατε την πρόσκληση, δεν υπάρχουν τροπολογίες για την ημερησία διάταξη. Ούτε υπάρχουν κάποιες ειδικέ ανακοινώσεις που θέλω να κάνω. Εκτός από ότι να σας πω ότι υπάρχει η μετάφραση των πρακτικών της περασμένης συνεδρίασης. έφτασε στα χέρια μας, υπάρχει στα... στο φάκελό σας. Το κύριο θέμα της ημερησίας διάταξης μας είναι να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς προβλέπουμε την εργασία στη δεύτερη φάση της εντολής μας και πώς θα διαμορφωθεί η τελική έκθεση. Το έχουμε συζητήσει έτσι στα σύντομα, όχι σε λεπτομέρειες όμως, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα και κυρίως γιατί πρέπει να θεωρήσουμε το εξής δεν μπορούμε να δεχθούμε χρονικές καθυστερήσεις όπως τις είχαμε στο πρώτο τμήμα των εργασιών μας. Δηλαδή, θα πρέπει να ψηφιστεί το θέμα αρχές Ιουλίου του επόμενου έτους στην Ολομέλεια. Αυτό σημαίνει, de facto, ότι θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει με την πρώτη διατύπωση του κειμένου της έκθεσης τον Μάρτι. Οτμάρ, ναι. Βρήκε τη σου. Ωραία. Επ' αυτού θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα στη συζήτηση. Πώς διαβλέπουμε την εργασία μας στο δεύτερο ημισή. Έχουμε την έκθεση όπως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια και αποστείλει στις 27 βουλές των κρατών μελών και έχουμε παρατήσει και μια σειρά ερωτήσεων τη συζήτηση και εξάρτηση των οποίων θεωρούμε σοβαρή. Και οι βουλευτές ταυτόχρονα ενημερώθηκαν ότι θέλουμε από κοινού τον επόμενο Μάρτιο να έχουμε μια συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες για να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και τι μπορούμε να έχουμε σαν τελικό αποτέλεσμα από την ανταλλαγή αυτή απόψεων και να δούμε ποια θα είναι ενδεχόμενα νομοθετικά μέτρα που θα μπορούμε να προετοιμάσουμε. Αυτά γενικά, τα ξέρετε. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας την Περβόν Περές να μας πει πώς βλέπει εκείνη τα πράγματα και μετά είσαστε όλοι καλόδεκτοι να συμβάλλετε στη συζήτηση. Παρακαλώ Περβόν. Merci, Monsieur le Président. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη συζήτηση που κάνουμε μετά από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Είναι σημαντική στιγμή και θα μπορέσουμε να προσανατολίσουμε τη συνέχεια των εργασιών μας σωστά. Θα έχουμε και μία συνάντηση των συντονιστών αμέσως μετά για να διευκρινίσουμε κάπως περισσότερο τα πρακτικά θέματα αλλά προς το παρόν σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δούμε πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα εδώ και ένα χρόνο, πώς πήγαν τα πράγματα στην Ολομέλεια και τι ε, προσανατολισμούς όπως είπα θέλουμε να δώσουμε. Πριν από την ψηφοφορία το μήνα Οκτώβριο, στις συζητήσεις που είχαμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων, είδαμε ότι υπήρχαν δύο σενάρια. Το πρώτο έλεγε ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε στις ερωτήσεις και η τελική έκθεση να είναι αυτή η οποία θα δίνει τις απαντήσεις. Ένα άλλο σενάριο είναι να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε για τις συστάσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε από αυτή τη φάση και ευτυχώς αυτό το δεύτερο σενάριο απεδείχθη εφικτό. Αυτό τι σημαίνει σημαίνει ότι στο μέλλον, στην επόμενη περίοδο μάλλον, η ουσία για μας είναι να γίνει μία προσπάθεια, θα έλεγα, εξυπηρέτησης των ιδεών και των συστάσεων τις οποίες προτείναμε στην Ολομέλεια και θα πρέπει όλες οι νομοθετικές προσπάθειες του Κοινοβουλίου από εδώ και πέρα να χαρακτηρίζονται από τις προτάσεις τις οποίες ήδη έχουμε περάσει στην Ολομέλεια. Βέβαια η κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ήδη από την πρώτη έκθεση και επιβεβαιώθηκε αυτό και από την ψήφο στην Ολομέλεια, η κρίση φαίνεται ότι συνεχίζεται. Ίσως επίσης να υπάρξουν και ορισμένες εξελίξεις ε, ε, στις οποίες θα πρέπει να επανέλθουμε, όπως το θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης της ζώνης ευρώ. Αλλά τα βασικά είναι στην έκθεση την οποία έχουμε περάσει. Και στα πλαίσια του, του χρονοδιαγράμματος το οποίο εσείς υποδείξατε θα πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή έτσι ώστε οι βασικές γραμμές της έκθεσης που ψηφίστηκε να χαρακτηρίζουν, να χρωματίζουν πλέον τα κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι βέβαια είναι σχετικό και θα είναι πολλά τα κείμενα αυτά τα έγγραφα αυτά. Τα θέματα τα οποία άπτονται της εκθέσεως της ειδική μας είναι πάρα πολλά βέβαια. Θα τεθούν και ορισμένα προβλήματα. Πρώτον, αναφερθήκατε στο θέμα του χρονοδιαγράμματος. Σημερίζομαι την εκτίμησή σας. Θελήσαμε να υπάρξει παράταση αυτής της εντολής για να συμπέσει με την διάρκεια της εντολής γύρω από την υπόθεση των δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό ε, νομίζω έχει μια κάποια λογική. Θα τα δούμε αυτά και στη συνάντηση των συντονιστών. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να οργανώσουμε ε, μία κοινή συνάντηση με την Επιτροπή Δημοσιονομικών Προοπτικών. Ξέρω ότι και αυτή έχει πάρα πολλή δουλειά και έχει πλημμυρίσει από θέματα και έχουν ξεκινήσει προς το σύνολο των κοινοβουλευτικών επιτροπών μια έκκληση ε, προς συνεργασία, προς ε, συνεισφορά των συγκεκριμένων ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών προς την Επιτροπή των Προοπτικών. Παρ' όλα αυτά πρέπει να οργανώσουμε αυτή την κοινή συνάντηση για να έχουμε μια πολιτική συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές, με τους πολιτικούς προσανατολισμούς που θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό. Δεύτερο, και σχετικά με τις συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες καλούμε να επεξεργαστούμε. Αν δεν συμβεί κάτι το ιδιαίτερο έκτακτο, η ουσία των προτάσεων ήταν ήδη στην πρώτη έκθεση. Και τέλος υπάρχουν το θέματα των σχέσεων με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Αυτό θα το συζητήσουμε σε επίπεδο συντονιστών νομίζω για να δούμε πρακτικά τι, τι γραμμή θα ακολουθήσουμε. Πάντως στα πλαίσια της ολομέλειάς μας αυτής εδώ, της Επιτροπής μας, να προσπαθήσουμε να δούμε ε, προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε σύμφωνα πάντα με αυτά που μέχρι τώρα έχουμε πετύχει. Ευχαριστώ, Περβόντς. Ήδη το Σεπτέμβριο ήρθα σε επαφή με την κυρία Χάου, που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής που αναφέρατε και οι δύο γραμματείες των Επιτροπών μας είναι σε συνεχή διάλογο. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή για την ε, οι δημοσιονομικέ προβλέψει δεν εργάζεται ακόμα, γιατί περιμένει να εγκριθεί ο προπολογισμό για το επόμενο έτο. Και έτσι η αρχική μα πρόθεση να έχουμε μια κοινή συνεδρίαση ήδη φέτο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το νωρίτερο το Γενάρη θα μπορέσουμε να συναντηθούμε. Έχουμε βέβαια εδώ μέλη που ανήκουν και στη, δική μας επιτροπή και στην Επιτροπή για τους Ο κύριος Σέγγιν έχει το λόγο. Ε, ναι, ε Πρόεδρε, για το θέμα αυτό, τα άλλα θα μπορούσαμε να τα εξετάσουμε αργότερα, όσον αφορά την Επιτροπή αυτή Τσούρ. Συμφωνώ με την εισηγητρία, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια κοινή συνεδρίαση. Όχι μόνο κοινή συνεδρίαση, αλλά να υπάρχουν και συντονισμοί μεταξύ των ΜΕΝ και των ΔΕ, γιατί πιστεύω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσουμε να βρούμε διέξοδο από την κρίση εάν δεν ε, τακτοποιήσουμε τον προπολογισμό μας. Είναι απαραίτητο αυτό. Δεν Θα ήθελα να προσεγγίσω προσοχή όμως ε, στο εξή, γιατί εγώ ανήκω και στις δύο επιτροπές. Ο εισηγητής Καρίγκα σκοπεύει τέλη Γενωρίου, άρχες Φεβρουαρίου, να υποβάλει στην Επιτροπή Τσούρε τους πρώτους του προσανατολισμού για τη τελική έκθεση. Και υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα μας αφορά γενικά, ε, το άλλο εμένα προσωπικά που πιστεύω ότι υπάρχουν θέματα που είναι σκανδαλώδη ότι δεν μπορούν οι εμπεριφερόμενες να δεχτούν ένα προπολογισμό που ξεπερνάει το 1% ας πούμε. Αυτό μου φαίνεται σκανδαλώδες. Τέλος πάντων. Το ένα αυτό το σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι εάν συμφωνήσετε με την κυρία Χάουκ ότι ίσως για να ίσως αργότερα συναντηθούμε και δύο μέρες αργότερα ο Σαλβατόρ υποβάλλει την, ε, το πρώτο προσχέδιο της έκθεσής του. Δεν θα μπορέσουν οι απόψεις να συμπεριληφθούν στα συμπαράσματα της Επιτροπής του. Θα ήθελα να επιτεσίσω την προσοχή σας στο θέμα αυτό, ότι πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα συντονισμός χρονικός. Και θέλω να υποστηρίξω την η συγγήτρια ότι θα πρέπει πραγματικά να εμπλακούμε με τη Ζούρε, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη και οι δικές μας απόψεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, τον Φρανκ Έγγελ και γιατί προτίθεται να βοηθήσει. Δεν ήταν δικό μας πάνω ορθής. Εμείς θέλαμε να υπάρχει συνάντηση αυτή και νωρίτερα. Αλλά ίσως με τη βοήθειά σου να το καταφέρουμε τελικά. Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα εκπρόσωπο του Σύνδεου Κοφεράτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω αντικαθιστώντας τον Κοφεράτη κάτι το οποίο ζήτησε και η κυρία Μπερές. Και έχει μεγάλη σημασία οι εργασίες μας, οι εργασίες της Επιτροπής μας να διεξαχθούν σε στενή σχέση με τους τομείς δραστηριότητας και με τις επιτροπές που εξετάζουν θέματα τα οποία όπως είπα άπτονται με παρεμβάσεις ε, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία να αναπτύξουν τη σχέση μας με την Επιτροπή ΣΟΥΡ, αλλά και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες σε αυτή τη βάση ασχολούνται με θέματα τα οποία, όπως είπα, ξανά συνδέονται άμεσα με την οικονομική κρίση και με τα υπόλοιπα επιμέρους θέματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση που έχει ήδη γίνει δεκτή για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, αυτά θα τα συζητήσουμε στο επίπεδο των συντονιστών. So, is... Ωραία. Όλοι ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω ένα πρακτικό θέμα. Το θέμα της συμμετοχής, της προσέλευσης των μελών στην Επιτροπή. Γιατί είναι δύσκολο να λέμε ότι εργαζόμαστε σκληρά, γιατί όντω το κάνουμε μερικοί, αλλά δεν συμμετέχει η ολόκληρη η Επιτροπή. Και για μένα αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και πριν επισέλθουμε στη συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος, ας σκεφτούμε πρώτα αυτό το θέμα της προσέλευσης. Ίσως δεν είναι εδώ η Επιτροπή κατάλληλη ευκαιρία, γιατί ελάχιστα τα μέλη ε, ελάχιστα μέλη βλέπω πέραν των συντονιστών, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το θίξουμε και αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, η συμμετοχή πράγματι και στο παρελθόν ήταν αρκετέ φορέ ανεπαρκέ. Αλλά βλέπουμε ότι όταν εμεί οργανώνουμε την εδρίασή μα πέμπτη απόγευμα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό, είναι δυστυχώ η παρουσία περιορισμένη. Γιατί πολλοί ήδη την πέμπτη το απόγευμα φεύγουν. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν όλα να συμμετάσχει στην ε, συνεδρίασή μας. Μπορούμε να κατονομάσουμε και να ντροπιάσουμε, να δημοσιάσουμε ένα κατάλογο ποιοι συμμετέχουν και ποιοι δεν συμμετέχουν. Αλλά τι να κάνουμε. Εγώ συμμερίζω με την απογοήτευσή σου, αλλά δεν βλέπω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση. Εκκλήσεις μπορούμε να προσθέσουμε. Στο παρελθόν οι εκκλήσεις αυτές δεν καρποφόρησαν. Και αυτό που με λυπεί είναι ότι ορισμένε πολιτικές ομάδες δεν εκπροσωπούνται καθόλου. Αυτό μου φαίνεται πραγματικό πολύ άσχημα. Οι πράσινοι παραδείγματος χάρη αρχής ε, δεν εκπροσωπούνται αρκετά παρόλο που έχουν και αντιπρόεδρο. Και αυτό πραγματικά δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. και το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά δεν θέλουν να στηρίξουν τα αποτελέσματα των εργασιών μας. Τίποτα άλλο επί του θέματος δεν έχεις να πεις. Για την εργασία στο δεύτερο ημισή. Όλε. Well, easier if more are here. Θα ήταν πιο εύκολο να ήμασταν περισσότεροι. Σίγουρα το κεντρικό θέμα για μας είναι η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, με τους εθνικούς βουλευτές. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ευρία συνένεση, και ευελπιστώ ότι θα το καταφέρουμε, τότε θα πρέπει να εμείνουμε στις συμβαστικές λύσεις. Ίσως να τις αξιολογήσουμε, να τις επεξεργαστούμε περαιτέρω αλλά να μην ανοίξουμε και πάλι το κουτί της Πανδώρας. Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Ας ε, διευκρινίσουμε ορισμένες πτυχές σε κάποια θέματα. Οι πράσινοι ήθελαν ε, να εξετάσουμε το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα, ενδεχομένως. Το ίδιο κάνει και η Οικονομική Επιτροπή. Αλλά προσοχή, προσοχή, να μην ξανανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Ρόπερ Τσίλε. Έχω να πω ότι μπορώ να συμφωνήσω με την Περβάνς Σπερέση. είναι σωστή αυτή η άγουσα ε, που μας οδήγησε στα αποτελέσματα των εργασιών μας στον πρώτο γύρο. Πετύχαμε συμβιβασμό και νομίζω ότι τη δεύτερη φάση αυτή θα πρέπει να είναι η βάση των εργασιών μας πάλι. Και θα ήθελα να προσθέσω αυτά που έγιναν ας πούμε επίκαιρα από τότε μέχρι σήμερα, αυτά που δεν εξετάσαμε πώς. Εγώ βλέπω κάποιες απόψεις τέτοιες. Καταρχήν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην έκθεση το θέμα του ιδιωτικού χρέους που αφορά και επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά στην Ευρώπη και τον συσχετισμό αυτών με διάφορα ταμεία ταμεία συνταξιοδότησης, cash flow, ε, κρατικό χρέος και τέτοια πράγματα που μπορούν να εξετάσουν στούν συγγνώμη περαιτέρω. Επίσης, οι ε, δημοσιονομικές προβλέψεις και η Επιτροπή των Δημοσιονομικών Προβλέψεων θα πρέπει να συντονιστεί μαζί μας, γιατί αν δεν συντονιστούμε και με την κοινωνική ε, συνοχή, θα οδηγηθούμε σε νέα βαθύτερη χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη. Άρα δεν θα έχουμε πετύχουμε κάτι καλό. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να παρουσιάσουμε πολύ συγκεκριμένε απόψει μα και τι ανησυχίε μα για την εξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την κρίση. Και τέλο, θα πρέπει επίση να σκεφτούμε τα εξή. Εγώ δεν είμαι μέλο τη Επιτροπή ΕΚΟ, τη Οικονομική Επιτροπή, εν αντιθέσει με πολλού που είναι εδώ, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει Αυτές οι έξι ε, νομικές πράξεις που εξετάζουν αυτή τη στιγμή στην Οικονομική Επιτροπή να εξαστεί και από εμά και νέα θεσμικά όργανα που δημιουργούνται λοιπά Και αυτό θα πρέπει να είναι σημαντικό για μας. Για τα άλλα θέματα θα εκφραστώ μέσα στα πλαίσια συνεδρίαση των συντονιστών. Και το θέμα της συνεργασίας με ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις των ε, βουλευτών πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Νικόλας Χούντης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή όπως είπατε κύριε Πρόεδρε και η συγγήτρια είναι η πρώτη συζήτησή μας μετά την ψήφιση της ενδιάμεσης έκθεσης στην Ολομέλεια και επειδή τώρα οργανώνουμε τη δουλειά μας στο επόμενο διάστημα θα ήθελα να κάνω ορισμένα γενικότερα σχόλια το πρώτο είναι ότι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. Είναι σωστή απόφαση που παρατάθηκε η, η εντολή μας για έναν ακόμα χρόνο. Το δεύτερο, όπως ξέρετε κύριε Πρόεδρε, με σεβασμό στις απόψεις που ακούστηκαν και στο τελικό αποτέλεσμα, την έκθεση την ενδιάμεση δεν την ψηφίσαμε. Και δεν την ψηφίσαμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους αναλύσαμε. Δεν θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα πρέπει να πάμε με την πρόθεση να μείνει αναλύωτη η έκθεση, διότι κατά τη γνώμη μας δεν είναι σωστή. Επομένως, η δική μας η προσπάθεια είναι να, η Επιτροπή μας να βγάλει στην τελική της έκθεση σωστότερα συμπεράσματα και να προτείνει σωστότερες προτάσεις. Αυτό θα είναι βεβαίως αντικείμενο του διαλόγου μας. Θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι συμφωνώ με όλες τις διαδικαστικές προτάσεις που έγιναν, να συνονοηθούμε, να συναντηθούμε, να κουβεντιάσουμε με άλλες επιτροπές, να προλάβουμε τις γενικότερες αλλαγές που γίνονται, αλλά αυτό που καταλαβαίνω σαν εντολή και σαν ευθύνη της Επιτροπής είναι πραγματικά να είναι εύστοχη όσο αφορά και τις αιτίες της κρίσης και το ξεπέρασμά της. Η εισηγήτρια σωστά είπε και είναι και η προσωπική μου γνώμη ότι η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί η σημερινή φάση της κρίσης, η φάση δημοσιονομική ή κρίση χρεών, σοβή, είναι σε εξέλιξη σε πολλές χώρες. Πολλά από τα μέτρα που λαμβάνονται και που δυστυχώς σε ορισμένα σημεία είναι μέσα στο πνεύμα της έκθεσης, γι' αυτό δεν την ψηφίσαμε, δημιουργούν οξύτερες καταστάσεις. Αν, κύριε Πρόεδρε, βάζαμε την έκθεσή μας σε ένα δημοψήφισμα στους ευρωπαϊκούς λαούς που σήμερα συναντούν σκληρά μέτρα στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στην Αγγλία, θα την απέρριπταν κατά τη γνώμη μου. Επομένω, η δική μα προσπάθεια πέρα από τι άλλε διαδικασίε θα πρέπει να είναι να εναρμονιστεί με τα αιτήματα για διαφορετικέ πολιτικέ, αναπτυξιακέ πολιτικέ στην Ευρώπη. Το λέω αυτό όχι για να πω ότι οι απόψει μου είναι σωστέ, αλλά γιατί πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα και η Επιτροπή μα πρέπει να δουλέψει πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα, πιο κοντά στι αγωνίε των Ευρωπαίων πολιτών. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε, δεν μπορούμε να δεσμευόμαστε από το τι θα πει η Κομισιόν. Άλλωστε, η Κομισιόν και η Σύνοδο Κορυφή ετοιμάζουν και λαμβάνουν μέτρα που αλλοιώνουν το θεσμικό οικοδόμημα τη Ευρώπη και ταυτόχρονα σκληρά μέτρα με τα πακέτα τη οικονομική διακυβέρνηση που κατά τη γνώμη μου δεν θα βγούμε από την κρίση και δεν θα βγούμε από την ύφεση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το σχόλιο ότι η δική μα προσπάθεια στη συνέχεια με τη συμμετοχή εδώ και τη συλλογική προσπάθεια είναι ε, να την κάνουμε καλύτερη την έκθεση. Και γι' αυτό θα συμμετέχουμε ενεργότατα και με τι προτάσει, σεβόμενοι και τι απόψει που θα ακουστούν. Πρακτικά τώρα, μια δεύτερη κατηγορία. Με βάση αυτέ τι σκέψει, ίσω στη συνάντηση των συντονιστών το κουβεντιάσουμε, έχω ορισμένε προτάσει και για τι επισκέψει σε χώρε. Θα τα πούμε ίσω μετά. Σα λέω, νομίζω ότι επιβάλλεται, επιβάλλεται επίσκεψη στην Ελλάδα είναι η πρώτη που εμφάνισε τα, όλα αυτά τα γρήγορα; Α, εντάξει, εντάξει. Ναι, λοιπόν, θα τα κάνουμε μετά και επίση ε, έχω και συγκεκριμένε προτάσει για αυτού που καλούμε εδώ και κουβεντιάζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε και ανθρώπου που τουλάχιστον ε, όταν οι άλλοι έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει κρίση, είχαν πει ορισμένα λόγια. Με αυτή την έννοια τη επιμέρου προτάσει αυτό, θα το συζητήσουμε μετά, ο Πρόεδρος. Αυτά τα θέματα που δείξατε στο τέλος θα τα συζητήσουμε μετά στους συντονιστές. Αλλά αναφερθήκατε σε ένα θέμα που είναι πολύ αμφιλεγόμενο κατά τη γνώμη μου. Εγώ το βλέπω διαφορετικό δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι η ουσία αυτό που θέλουμε να πούμε και το εκφράσαμε στην ενδιάμεση έκθεση θα πρέπει να αμφισβητηθεί, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Κατ' εμέ, το αποτέλεσμα που ψηφίσαμε μέχρι στιγμή, στο Σεπτέμβριο δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής μας. Και ήταν ένα αποτέλεσμα στο οποίο φτάσαμε μετά από σκληρέ προσπάθειες. Και είναι και ένα αποτέλεσμα που αποτελεί ένα συμβιβασμό. Καμία πολιτική ομάδα δεν ικανοποιήθηκε 100%. Γενικά όμως αυτός ο συμβιβασμός θεωρήθηκε αποδεκτός. Εάν τώρα ξανανοίξουμε το κουτί της Περδόρας και πούμε ότι θέλουμε να έχουμε νέα συμπεράσματα, δεν θα ήταν κάτι που θα με έβρισκε εμένα προσωπικά σύμφωνο και δεν ξέρω αν η πλειοψηφία της Επιτροπής θα το ήθελε. Δεν θα συνιστούσα να ακολουθήσουμε την άγουσα αυτή. Στον Βασβάγγελ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι ένα από τα μέλη της Επιτροπής για την κρίση που δεν είναι οικονομολόγος, δεν έχει τέτοιες γνώσεις. Παρακολούθησα το πρόγραμμα αυτής της Επιτροπής και υπό ένα άλλο πρίσμα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα χρηματοπιστωτικά μέσα και την οικονομική διακυβέρνηση. Όπως είπε και ο προλαλής σας συνάδελφος από την Ελλάδα, η κρίση έχει πολύ διαφορετικές ρίζες και αντιμετωπίστηκε με πολύ διαφορετικό τρόπο στις χώρες. Και παρόλο που δεν είμαι οικονομολόγος, πιστεύω ότι μέχρι στιγμής το έργο αυτής της Επιτροπής ήταν εξαιρετικό και επέφερε και προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι είχαμε την αφρόκρεμα της οικονομικής ε, γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης μέχρι στιγμής. Ίσως όμως στις επόμενες φάσεις στο μέλλον να προσκαλέσουμε ανθρώπους, όχι κατά ανάγκη εμπειρογνώμονες, ανθρώπους που προβληματίζονται για τις ρίζες της κρίσης υπό άλλο όμως πρίσμα, όχι υπό το αμυγός οικονομικό. Νομίζω ότι έτσι θα εμπλουτίσουμε τη συζήτησή μας, αν ξεπεράσουμε το οικονομικό περίσμα. Επίσης, ε, καλό θα ήταν να αναμίξουμε και τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών. Να ρωτήσουμε τους εθνικούς βουλευτές τι έκαναν το χρόνο που πέρασε, τι έκαναν από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Γιατί συμφωνήσαμε για κάποιες κοινές, για κάποια κοινά μέτρα και κοινό τρόπο αντιμετώπισης σε επίπεδο Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, αλλά υπήρξαν και ειδικά μέτρα και πολύ συγκεκριμένες αντιδράσεις που υιοθετήθηκαν από μεμονωμένες χώρες και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τις ιδιαίτερες αυτές προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης. Να δούμε λοιπόν τι έγινε τελευταία σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές χώρες της Ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ευχαριστώ. Έχω τώρα την Ουγγαρέζα συνάδελφα μα, έχει το λόγο. Úr, ε, nagyra értékelem a jelentést, és nagyon fontosnak tartom minden megállapítását. Később kapcsolódtam be új képviselőként a bizottság. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είμαστε, είμαι καινούρια στι εργασίε εδώ τη Επιτροπή. Θεωρώ όμω η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή και είναι καλή βάση για τι μελλοντικέ εργασίε. Όσον αφορά την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε, εγώ θα υποστήριζα την συνένεση και συνεργασία, όπω ανέφερε και η συγγήτρια. Όλοι οι εμπειρογνώμονε των οικονομικών συμφωνούν ότι δεν έχει λήξει ακόμα η κρίση και ότι η κρίση θα μπορεί να επαναληφθεί εκτό αυτού. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη που έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν ή να αποφύγουν την κρίση και έχουν αποκτήσει κάποιες γνώσεις, θα πρέπει αυτές οι γνώσεις να ληφθούν υπόψη ε, για τη μελλοντική μας εργασία. Να ξέρουμε τις πρακτικές αυτές και θα πρέπει να κάνουμε μια αναθεώρηση να δούμε τι δεν έχει εξεταστεί, τι έχει αφαιθεί κατά μέρος και τι οδήγησε στην κρίση. Το τρίτο, ποια θα είναι η μέθοδος για την συνόδευση και ανάλυση της κρίσης. Η συνεργασία μια σειρά σε επιτροπών ασχολούνται με το θέμα αυτό. παραδείγματο χάρη ένα πρόγραμμα ε, της ανά, ανάλυσης των δικτών που εκτός από το ΑΕΠ μπορούν να ληφθούν υπόψη για να υπάρχει μια προειδοποίηση για επικείμενη κρίση. Η επόμενη παρατηρήση αφορά το εξή. Μια που δεν θα δούμε το σημείο στο οποίο τελειώνει η κρίση, και θα πρέπει από την άλλη μεριά να δούμε πώς θα εκτιμήσουμε την κρίση αυτή και είναι πολύπλοκο το θέμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίζουμε τις εργασίες μας και αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη παρατήρηση από αυτού. Γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Από όσοι κατάλαβα εγώ, εργαστήκαμε πάρα πολύ έντονα πάνω στο θέμα των αιτιών της κρίσης. Και μια συμπληρωματική ανάλυση ίσως θα δώσει κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, αλλά μόνο πολύ μικρά και όχι τεράστια σημασίας. Γιατί την ανάλυση την κάναμε πραγματικά εις βάθος και την αξιολόγηση επίσης. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις βέβαια, αυτό εξαρτάται και από την πολιτική, τον πολιτικό προσανατολισμό. Ο ένας θεωρεί αυτός ο παράγοντας είναι πιο σημαντικός, ο άλλος θεωρεί ο άλλος είναι πιο σημαντικός. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε πολλά εάν τώρα ξαναρχίσουμε να εξετάζουμε τα αίτια. Όσον αφορά την επιτήρηση, αυτό είναι ένα θέμα που εξετάσαμε επίσης αναλυτικότατα και από την Αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. και συμφωνήσαμε να υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή αρχιδομή αν θέλετε επιτήρησης και θέλω να σας υπενθυμίσω το εξή. Έχουμε λίγο χρόνο αυτή τη φορά. Σε 5-6 εβδομάδες είναι Χριστούγεννα, μέχρι τότε δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα και θα αρχίσουμε μετά στις 10 Ιανουαρίου. Και μέσα Μαρτίου θα έπρεπε να έχουμε το τελικό έγγραφο. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε ρεαλιστές. Θα είναι δύσκολο τα εθνικά κοινοβούλια που μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, τα εθνικά κοινοβούλια λέω να εμπλακούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να μπορούμε να πούμε αυτή είναι μια έκθεση την οποία έχουν δεχθεί όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι ο κύριο μας στόχος. Τώρα να προσποιηθούμε ότι έχουμε απεριόριστο χρόνο για να κάνουμε χιλιάδε αναλύσει δεν είναι σωστό, δεν έχουμε τον χρόνο αυτό και οπωσδήποτε θα θέλω να αποφύγω του χρόνου να ξαναζήσουμε αυτό που είδαμε στην αρχή που δεν ήσασταν εσείς εδώ που ο χρόνος μας έλειπε και αναγκάσαμε να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφο Τανούτα Χούμπνερ. Uh, Σας ευχαριστώ. Λυπούμε, αλλά δεν παρακολούθησα τη συζήτηση από την αρχή και ίσως πω κάτι αντιφατικό ή επαναληπτικό, αλλά θα ήθελα να κάνω παρόλα αυτά δύο-τρία σχόλια. το γεγονός ότι οι συστάσεις και η οριστική έκθεση με τις συστάσεις θα εγκριθούν γύρω στον Ιούνιο δικαιολογούν την ανάγκη να είμαστε πιο ευρύ στις συστάσεις μας, δηλαδή να μην περιοριστούμε στην κρίση, να δώσουμε πιο διευρυμένο περιεχόμενο. Θα αντιλήσουμε βέβαια κάποια συμπεράσματα από την ανάλυση των ε, αιτίων της κρίσης και θα μιλήσουμε για την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων, αλλά ήδη θα έχουν ξεκινήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις, όπως αυτή των χρηματοπιστωτικών αγορών ή θα ετοιμάζονται όπως αυτή της οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να περιοριστούμε σε τέτοιες μόνο συστάσεις. Θα πρέπει να είμαστε και πιο διορατικοί, να θετήσουμε ένα πιο μακροπρόθεσμο πρίσμα, γιατί πολλές από τις συνέπειες της κρίσης θα τις βιώσουμε στο μέλλον. Γιατί δεν έχουμε μόνο ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης, η κρίση είναι παγκόσμια. Οπότε, σε αντίθεση με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η δική μας ευθύνη είναι να κοιτάξουμε το σφαιρικό πλαίσιο, την παγκόσμια οικονομία και φυσικά και το ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Αλλά στις συστάσεις μας θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένες πτυχές ε, της ανάλυσης των αιτίων, αλλά που δεν αναπτύσσονται περαιτέρω στις μεταρρυθμίσεις ή στην κοινοτική νομοθεσία. Επειδή ακριβώς ε, δεν εμπίπτουν στις κοινοτικές αρμοδιότητες. Το καθήκον μας λοιπόν θα ήταν μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου που θα κορυφωθεί η συζήτηση για την έκθεση να υιοθετήσουμε συστάσεις που θα είναι πιο διορατικές και θα υιοθετήσουν πιο φιλόδοξο χρονικό ορίζοντα. Δεν θα περιορίζονται στις μεταρρυθμίσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, συμφωνώ μαζί σας ότι η ανάλυση έγινε, μπορεί να μην ήταν ιδεώδης, αλλά οι αναλύσεις τέτοιου είδους κρίσεων ε, θα είναι μακροχρόνια. Το ίδιο συνέβη και με την κρίση του... με προηγούμενες κρίσεις που χρειάστηκαν 20 και 30 χρόνια για να ερμηνευθούν. Είναι πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα της ανάλυσης. Οπότε συμφωνώ να μην ε, επαναλάβουμε τη συζήτηση, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρούμε αυτή την ανάλυση ως κάτι ε, απαράβατο και ιερό για τη συνέχιση της συζήτησης θα βελτιώσει και την ποιότητα της ενδιάμεσης μας έκθεσης. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας να μην ξαναρχίσουμε τη συζήτηση που έγινε, αλλά αν υπάρχει καμιά καλύτερη πρόταση θα πρέπει να την απορρίψουμε μόνο και μόνο για να μην ξαναρχίσουμε τη συζήτηση. Σε ό,τι φορά το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης, Κατά τη γνώμη μου είναι καθήκον μας να πραγματοποιήσουμε την πρώτη αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα του συνόλου των μεταρρυθμίσεων γιατί έχουμε τις διάφορες επιτροπές που ασχολούνται με συγκεκριμένες πτυχές ορισμένες επιτροπές για τις χρηματοπιστωτικές αγορές μια άλλη επιτροπή για την εσωτερική αγορά μια επιτροπή για την εξωτερική εκπροσώπηση αλλά εναπόκειται σε εμά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. για το σύνολο των μεταρρυθμίσεων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να οργανώσουμε μία ευρεία συζήτηση. Όχι όμως μία συζήτηση όπως γίνεται στο Κοινοβούλιο για τις τροπολογίες ε, της έκθεσης και την εγκαλότητα Κόλλα, μια γενικότερη συζήτηση για την κρίση, για την Ευρώπη που εξέρχεται από την κρίση. Μία συνδιάσκεψη υπό την αιγύδα της δικής μας Επιτροπής που θα αξιολογήσει τις μεταρρυθμίσεις και θα προτείνει τρόπους για μελλοντική δράση. Και εκεί ίσως θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και την έκθεση Ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει μια αρχική αξιολόγηση του συνόλου των μεταρρυθμίσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ αποσπασματική και κατακαιρματισμένη η ανάλυση αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και για τα Εθνικά Κοινοβούλια αντιλαμβάνουμε τη σημασία της ε, επαφής, αλλά είναι πολύ δύσκολο και όλες οι συνεδριάσεις που είχαμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια τον τελευταίο χρόνο και εμπειρία μου από την πιο πρόσφατη συνάντηση είναι ότι κάτι πάει στραβά. Δεν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αυτή την κρίσιμη μάζα της ανταλλαγής απόψεων, να βρεθούμε στο ίδιο μήκος κύματος. Οπότε έχουμε προγραμματίσει από ό,τι βλέπω για το Μάρτιο συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά καλό θα ήταν να προετοιμάσουμε αυτούς τους συναδέλφους ε, που θα έρθουν από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να μπορούν να είναι κατατοπισμένοι όταν συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάτι που δεν συνέβη στο παρελθόν, τουλάχιστον από τις συνεδριάσεις που είχα εγώ εμπειρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντανίτα Βίμπνερ. Στο τελευταίο σημείο έχετε μαζί πείτε τα δίκαια. Η συμμετοχή και η προετοιμασία των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν ήταν πάντα ικανοποιητική και δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε βελτίωση. Μου φαίνεται καλή ενδιαφέρουσα η πρότασή σας ότι θα μπορούσε ίσως η Κομισιόν να οργανώσει μια μεγαλύτερη εκδήλωση για να δούμε κατά πόσο βάση των αναλύσεων που έχουμε ήδη δεν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε κάποιες προτάσεις μας. Ιδίως όσον αφορά τα μελλοντικά χρόνια τη εξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να το εμφαθύνουμε τόσο στη συζήτηση. Οι εκθέσει έχουν ζητήσει το λόγο. Äh, Α, τελευταία. Ωραία. Εισηγήτρια στο τέλο. Νομίζω ότι η ανάλυση ακούστηκε ήδη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία αναλυτικά στην ίδια την ενδιάμεση έκθεση. Δεν είναι καινούργια όλα αυτά γιατί έτσι και αλλιώ πάρα πολλοί εμπειρογνώμονες πολιτικοί ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά πριν εμείς κλείσουμε αν θέλετε με την ενδιάμεση έκθεση. Και όποιος θέλει να διαβάσει υλικό μπορεί να διαβάσει χιλιάδες σελίδες για το σύνολο των θεμάτων τα οποία οδήγησαν στην κρίση αυτή. Μόνο για την Ισλανδία στη βιβλιοθήκη μας υπάρχουν 2.000 σελίδες για να δείτε δηλαδή ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε νέα ανάλυση. Το εύρος της ανάλυσης επίσης έχει μεγάλη σημασία. Τώρα πρέπει να εμβαθύνουμε. Τα στοιχεία υπάρχουν στην ενδιάμεση έκθεση σε εμβριακή ίσως κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά ε, δεν χρειάζεται, όπως είπα, να βρούμε καινούργια πράγματα. Η ενδιάμεση έκθεση αυτή νομίζω είναι τμήμα των συμπερασμάτων μας, είναι ένα πρώτο εισαγωγικό τμήμα, είναι η βάση του δεύτερου ημίσεως των εργασιών μας και δεν χρειάζεται βέβαια να επανέλθουμε σε θέματα στα οποία έχουμε ήδη ψηφίσει, έτσι δεν είναι αλλά σε θέματα τα οποία είναι ακόμα προσυζήτηση. Και να πω επίσης ότι έχω βαρεθεί, μα έχω βαρεθεί με τις ακροάσεις. Δεν θέλω να συναντήσω κανένα εμπειρογνώμονα, βαρέθηκα. Τους ακούσαμε όλους. Ακούσαμε ακόμα και ανθρώπους που δεν ήταν εμπειρογνώμονες και τους κάναμε εμπειρογνώμονες μόνο και μόνο για να τους ακούσουμε. Λοιπόν, μιλήσαμε πολύ για εποπτεία, για έλεγχο και αν κάτι κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ακριβώς εποπτεία και έλεγχος και όλη η Ευρώπη βέβαια, είναι το μόνο που κάναμε. Αυτό που με θλίβει είναι ότι εδώ και δύο χρόνια συνειδητοποιούμε το τι συμβαίνει. Και το μόνο που κάνουμε είναι να ελέγχουμε την κατάσταση, να έχουμε μια εποπτεία της κατάστασης. Έγινε αυτό, το κάνουμε αν δεν έγινε και δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε τη συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Η συζήτηση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τώρα πρέπει να φτάσουμε, θα έλεγα, στο πολιτικό κομμάτι. Ο έλεγχος και η εποπτεία με ό,τι αυτό... Πολιτικό, με ό,τι αυτό σημαίνει είναι δύσκολο να δούμε πώς θα τα οργανώσουμε, πώς θα συνδέσουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο εποπτείας με τα εθνικά επίπεδα. Είπαμε ότι οποιοδήποτε δημοσιονομικό, ε, συγγνώμη, χρηματοπιστωτικό προϊόν σε όλο τον κόσμο δεν θα πρέπει να διαφεύγει ασδήποτε μορφή ελέγχου. Ωραία, εντάξει, το είπαμε σε επίπεδο αρχής, πρέπει να είμαστε βέβαιοι και πώς θα το πετύχουμε. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία όμως τα οποία με απασχολούν. Το πρώτο είναι το δημόσιο χρέος. Και τι συνέπειες έχει το δημόσιο χρέος. Θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι οι οποίοι απειλούν αυτή τη στιγμή την Ήπειρό μας. Κάποιοι από τους κινδύνους αυτούς είναι εσωτερικής παραγωγής, κάποιοι άλλοι είναι εισαγόμενοι. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό χωρίς ιδεολογία. Το να λέμε ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε την οικονομία είναι κάτι το οποίο το έχουμε βαρεθεί. Ο Κέινς δεν θα μας το έλεγε αυτό πια γιατί ιδιαίτερα στη λογική του Κέινς παρόλα αυτά παράγουμε θα έλεγα πλεόνασμα και όχι απλά δεν κινητοποιούμε απλά την παραγωγή, δεν αυξάνουμε απλά την παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν ας ξεφύγουμε από αυτή τη λογική. Σχετικά τώρα με τις ανισότητες στο διεθνές εμπόριο, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι Ευρωπαίοι γύρω από το θέμα των ανισοτήτων των εμπορικών και κάποιες άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία, η Ινδονησία κτλ. Και όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τις ισοτιμίες των νομισμάτων στο μέλλον και την νομισματική πολιτική. Και εδώ από ό,τι φαίνεται ξεσπάει ένας καινούριο πόλεμος. Σήμερα το πρωί φαίνεται ότι σε σχέση με αυτό το αυτή την εξαιρετική δήλωση την οποία κάναμε, ψήφισμα που κάναμε, προσθέσαμε πολλές σελίδες υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ μας κήρυξαν τον πόλεμο πριν μια εβδομάδα. Και το κίνιο βούλιο μας και ίσως και το σύνολο της Υπήρου δεν το πήραν είδηση. 600 δις δολάρια αντί να τροφοδοτούν την Αμερικανική οικονομία γιατί αν το έκαναν αυτό τα ποσά αυτά που είχε ήδη έτσι γίνει με τα 380 εκατομμύρια δις μάλλον τα οποία έχουν διατεθεί, δημιουργούν προβλήματα στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι λοιπόν μείζον το πρόβλημα, τίθεται το θέμα των μέσων της νομισματικής πολιτικής που θα πρέπει να έχουμε στην Ευρώπη, τον ρόλο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, η οποία σε κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να παρέμβει στον τομέα των ισοτιμιών. Μπορεί να ξαναβρεθούμε τους επόμενους μήνες ή χρόνια σε μια κατάσταση διαχείρισης του ύψους του ευρώ. Ε, μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν θεωρούσαμε ότι μπορεί να συμβεί, αλλά επί της ουσίας αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο και πρέπει να το συζητήσουμε και να μην κάνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται διότι είναι αιρετικό. Και τελευταίο θέμα, το συζητήσαμε και διμερός και πολυμερός, πρέπει να κλείσουμε σχετικά με τα συμπεράσματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την πολιτική Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν έχουμε φτάσει πουθενά σε σχέση με τα πολιτικά συμπεράσματα της κρίσης. Συντονίσαμε, εποπτεύουμε, ελέγχουμε, αλλά τελικά εξακολουθούμε να έχουμε πολλούς ε, ε, εμπλεκομένους, ενώ θα έπρεπε να έχουμε κατά περίπτωση ένα και εδώ έρχεται η πρόταση της Περβάνς σχετικά με τον συντονισμό των αρχών που ασχολούνται με τα θέματα της εποπτείας. Πρέπει λοιπόν να τα συζητήσουμε και αυτά τα πολιτικά συμπεράσματα. Γι' αυτό λοιπόν, λέει και ο Σέγγελ, τους επόμενους μήνες θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις ανάμεσά μας, σημαντικές συζητήσεις, όλα τα στοιχεία τα έχουμε και θα πρέπει να συμφωνήσουμε στις πολιτικές προτάσεις γιατί την πολιτική ε, είναι αυτή που μας λείπει και όχι η εμπειρογνωμοσύνη. Ευχαριστώ για τις σαφείς αυτές δηλώσεις και κάπως προκλητικά λόγια που παρουσιάσετε που εν μέρη συμμερίζομαι, όχι πλήρως, αλλά εν μέρη. Και πραγματικά η εξελίξη των τελευταίων ημερών θα έπρεπε να μας κάνουν και εμάς να εξετάσουμε το ένα το άλλο θέμα μπορούμε να το ενδεβαθύνουμε συνεδρία των συνεδριστών. Κύριε Απέτη Κάνεν, να πάρει το λόγο και μετά υπερβάσω. Thank you very much. I'm sorry for... Ευχαριστώ. Λυπάμαι που καθυστέρησα, αλλά είχα και άλλη συνεδρίαση. Θα είμαι λακωνική όπως το συνηθίζω. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι καλό θα ήταν να μην ξανανοίξουμε τη συζήτηση και την έκθεση, να μην αναδιατυπώσουμε την ανάλυση, να μην αμφισβητήσουμε την ανάλυση για τις ρίζες και τα αίτια της κρίσης. Επίσης, συμφωνώ με τις προοπτικές και συμφωνούμε να υιοθετήσουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και να είμαστε πιο διορατικοί. Επίσης, θα ήταν συνετό να αξιολογήσουμε το κατά πόσο οι μέχρι τώρα αποφάσεις ήταν χρήσιμες για την οικονομία. Και επίσης ε, να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ποιες ήταν οι ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικές στην παγκόσμια οικονομία. Και αντί να έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο προτάσεων και δημοσίων ακροάσεων, καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά ζητήματα. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Δεν είναι εξαντλητικός ο κατάλογος. Σε ό,τι αφορά την ε, ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. δεν ξέρω αν θα πρέπει να έχουμε μια έστω και κλεισμένη το θηρόν συνάντηση με τον Όλη Ρένι και άλλους επιτρόπους για να δούμε ποια θα είναι τα μελλοντικά μας βήματα για το δημόσιο χρέος ή για την ευθυγράμμιση των εθνικών προπολογισμών. Υπάρχει διαφορά σε ό,τι αφορά την ε, φορολογική πολιτική μεταξύ της Ευρώπης και των υπόλοιπων εταίρων. Για την ε, ρύθμιση, για τους κανονισμούς, καλό θα ήταν να έχουμε μια συνάντηση και με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Επίσης, να δούμε τι μπορούμε να πούμε ε, για την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, για, γιατί η μεταρρύθμιση του Διεθνούς Μεσματικού Ταμείου δεν ήταν αυτή που περιμέναμε και η G20 είναι τελείως αναποτελεσματική συνάντηση και έχει γίνει περίγελος. Υπάρχουν όμως τόσο τεράστιες διαφορές στην αντιμετώπιση φορολογική και δημοσιονομική πολιτική και καταλαβαίνω γιατί είπα λαμβάνουν τα μέτρα που λαμβάνουν και γιατί η Κίνα υιοθετεί τη δική τη πολιτική. Το θέμα είναι εμεί τι κάνουμε. Τι να κάνουμε, να, να υποτιμήσουμε το νόμισμα είναι ίσως λογικό, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αποτελεσματικό για οποιονδήποτε. Το θέμα είναι τις διάφορες δομές λήψης αποφάσεων για τη φορολογική πολιτική, πώς θα καταφέρουμε να τις συνδυάσουμε. Μία τέτοια συζήτηση είναι απαραίτητη. Ό,τι αφορά την φορολογική και δημοσιονομική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική πολιτική. Θα μπορούσαμε για την επόμενη μεταρρύθμιση να έχουμε ένα είδος έκθεση τελαροσιά για την πράσινη οικονομία. Η επόμενη μεταρρύθμιση του IFRS. να εκτιμήσουμε την αξία των σημάτων και της εικόνας των ε, επιχειρήσεων ή να δούμε τους λογιστικούς κανόνες. Επίσης, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα των πόρων, η επίπτωση στις κλιματικές αλλαγές. Δεν είναι ξεχωριστά θέματα αυτά από την οικονομία. Παρόλο που αυτή τη στιγμή διαχωρίζονται. Επίσης, τα νέα και νοτόμα προϊόντα που συνέχεια παράγονται. Να έχουμε μια γενική αρχή διαφάνειας. Γιατί μπορεί να είναι καλά τα νέα προϊόντα, αλλά θα πρέπει να ισχύουν παντού οι ίδιοι κανόνες, να υπάρχει διαφάνεια. Και μία προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική το 2020. Και καλό θα είναι να, να συντονίσουμε την πρότασή μας με την ε, Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά να μην εξετάσουμε μόνο τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η, η διάρθρωση της ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ε, για την καινοτομία. Τι γίνεται, τι γίνεται με τις συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει να επενδύσουμε προγράμματα που είναι πολλά υποσχόμενα για το μέλλον και αυτό δεν γίνεται μέχρι στιγμής, δεν γίνεται αρκετή συζήτηση. Αυτό θα ήταν, μια και περιμένουμε τα Χριστούγεννα, αυτό θα ήταν το γράμμα προς τον Άγιο Βασίλη και λέω ναι στη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτές τις συνεδριάσεις, γιατί να μην ζητήσουμε και από τα Εθνικά Κοινοβούλια να συστήσουν δικές τους επιτροπές προβληματισμού και να μας στείλουν ε, τις εκθέσεις τους. Γιατί αυτές οι συζητήσεις που γίνονται δεν είναι και πολύ παραγωγικές. Κοιτάξτε, ενημερώθηκαμε πώ εξετάζουν την κρίση τα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχουν ορισμένε χώρε που έχουν μια δική του επιτροπή κρίση. Έχουμε τον συνάδελφο εδώ από τι κάτω χώρε, κ. Στο Βέλγιο υπάρχει μια τέτοια επιτροπή, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία, ορισμένε χώρε που δεν έχουν ίσω επίσημη επιτροπή κρίση, αλλά έχουν κάποιο είδο τέλο πάντων ανεπίσημη επιτροπή. και πρέπει εκείνοι να κρίνουν κατά πόσο θέλουν ή δεν θέλουν να έχουν μια επιτροπή. Εγώ νομίζω ότι έχουμε κάθε συμφέρον να έχουμε τις δικές τους αντιδράσεις. θα πρέπει να προσπαθήσουμε ιδίω όταν υποβάλλουμε τέτοιου είδους ε, προτάσεις όπως τις ε, προτείνει ο Φρανκ Έγγελ, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς τη συμφωνή γνώμη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί σύμφωνα και με τις Ειδίκες Λισαβόνας, έχουν οπωσδήποτε δικαίωμα λόγου. Και αν έχουν την εντύπωση ότι τα δικαιώματα τους επικουρικότητας πλήττονται, θα είναι πάρα πολύ κακό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι γιατί πολύ μου κάτι δεν κάνουμε. Υπερβώς. Α, όχι, συγγνώμη. Και εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί δεν παρακολούθησα από την αρχή τη συζήτηση. Πάντως νομίζω ότι το έργο που επιτελέσαμε στην πρώτη φάση ήταν σημαντικό και θα μπορούσαμε στη συνέχεια να ασχοληθούμε και με το θέμα της αηφορίας ή μερισμένα πράγματα που απασχόλησαν και το G20. Για παράδειγμα, το συνολικό ε, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πώς λειτουργεί, ποια θα είναι η μελλοντική του διοργάνωση, ποια αρχιτεκτονική θα πρέπει να έχει αυτό το σύστημα. Ποιος είναι ο ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Επιτροπή της Βασιλείας. Πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά στη, στη δική μας αρχιτεκτονική των θεσμικών οργάνων. Τι θα γίνει με τις άλλες δικαιοδοσίες. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και θα αποτελέσουν τμήμα της μελλοντική μας ανάλυσης και προβληματισμού. Υπάρχει και ένα άλλο γενικό θέμα που είναι πολύ σημαντικό αφορά την μακροοικονομική διεθνή συνεργασία. Αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας, αλλά και του Παγκόσμιου Προγράμματος Εργασίας. Υπάρχουν ανισορροπίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχουν ανισορροπίες και παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός χρηματοπιστωτικός χώρος σε ολόκληρο τον κόσμο, οπότε έχουμε μεγάλες ευθύνες και αν δεν λάβουμε τις σωστές αποφάσεις θα χάσουμε βάρος, ειδικό στο μέλλον. Είναι σημαντικό να γίνει μια τέτοια ανάλυση λοιπόν με διορατικότητα. Μετά την αποτυχία των θεσμών του Bretton Woods είχαμε πολλές κρίσεις, ε, οικονομική, νομισματική, χρηματοπιστωτική, αδυναμία πληρωμών. Ποιες είναι οι προοπτικές του Διεθνούς ε, Νομισματικού Συστήματος και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης για τα θέματα, τα κανονιστικά και τις ρυθμίσεις, μην ξεχνούμε και τα θέματα τα φορολογικά. Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών επίσης είναι σημαντικό ζήτημα. Και το θέμα της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτή η κρίση ξεκίνησε από τα subprime, έγινε χρηματοπιστωτική, επηρέασε τα οικονομικά των κρατών μελών και υπονομεύει την ίδια μας την ανάπτυξη. Θα πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε λοιπόν την οικονομία και να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα της οικονομικής διακυβέρνησης που παρατηρούμε παγκοσμίω. Δεν θα πρέπει να περιορίσουμε την ανάλυση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το δούμε παγκοσμίω. Τι γίνεται με το G20, ποιες είναι οι προπτικές. Το παγκόσμιο πλαίσιο υπό το πρίσμα και των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα αναλύσουμε στη δεύτερη φάση και επαναλαμβάνω εκ παραλλήλου με τα ζητήματα που αναλύει η G20. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Ίσως να επανέλθω σε κάποια από αυτά που ακούστηκαν στη συζήτηση. Καταρχάς κάτι που ξέχασα εγώ ίδια να πω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε, γιατί δεν ήταν προφανές εξ αρχής ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αυτό το ευτυχές σενάριο χωρίς να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Νομίζω ότι αυτή ήταν ε, η προσπάθεια αποτέλεσμα της συλλογική συνειδητοποίησης του μεγέθου της κρίσης. Δεν ξέρω επίσης αν ε, συμμερίζεστε την δυσθυμία μου στο συγκεκριμένο τομέα είναι λογικό να εξετάζεται η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια σαν στρατηγικής φύσεως συζήτηση την Τετάρτη. Αλλά η σύγχυση με την προπαρασκευή της ομάδας των 20 και του Συμβουλίου και την έκθεση ΦΕΟ νομίζω ότι δεν ήταν πολύ καλή ιδέα. Δημιουργήθηκε κάποια μορφή παρανόησης. Οι υπόλοιπε συζητήσει συγκεντρώνονται σε θέματα μικροπρόθεσμα, θα έλεγα βραχυπρόθεσμα, συγγνώμη, και ε, χάνουμε την προοπτική που απαιτείται για, τις δικές μας, για τη δική μας προσπάθεια. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στο δεύτερο κομμάτι της έκθεσης. Κάτι το οποίο παρέλειψε επίσης να πω είναι ότι στο, στο ιδιαίτερα ε, ε, στενόχρονο διάγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουμε να δούμε τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή αυτή η ειδική για τις προοπτικές τη μελλοντική χρηματοδότησης κτλ. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ζητήσαμε την παράταση λειτουργίας ήταν η αισιόδοξη αν θέλετε άποψη την οποία έχουμε ότι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και αυτό το αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε από κοινού δυσκολευόμαστε σε εισαγωγικά να το πλασάρουμε. Τι λέμε εδώ και συμφωνώ με τον συνάδελφο Έγγελς. Λέμε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να ξυπνήσει, να καταλάβει ότι έχει κάτι να πει, ότι έχει κάτι να προασπιστεί και το θέμα είναι ακριβώς να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις συγκεκριμένες αυτές προτάσεις κάτω από τους γνωστούς περιορισμούς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουμε ή όχι την χρηματοδότηση. Για τις αιτίε. αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις αιτίε ίσως και να έχουν δίκιο. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο δυσκολευόμαστε να συμφωνήσουμε. Υπάρχει μια αντίφαση όμως εδώ. Κάποιοι με κατηγόρησαν να επιβαρύνω το σκάφος εις βάρος των χρηματαγορών. Από την άλλη, στην πραγματικότητα, δούμε τις αιτίε οι οποίες είναι ανιχνεύσιμες έχουν σχέση ακριβώς με την λειτουργία των χρηματαγορών. Εγώ θα ήθελα και πιο βαθύτερες αιτίε ή αναλύσεις για πιο βαθύτερες αιτίες. αιτίες που έχουν σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες σαν παράδειγμα. Αν λοιπόν θεωρήσουμε σε κάποια φάση ότι στα πλαίσια της Επιτροπής μας υπό το φως του τι θα ακολουθήσει υπάρχει μια κάποια συνένεση η οποία θα λέει ότι πράγματι η κοινωνική ανισότητα τροφοδότησε τις αιτίες αυτής της κρίσης. Αλλά θα το πούμε αυτό όταν βλέπω τι γίνεται στο Συμβούλιο και όταν βλέπω τι γίνεται γύρω από μας, δεν βλέπω να επιμένει κανείς γύρω από αυτό το θέμα και δεν ξέρω τι θα κερδίσουμε εμείς αν το ανοίξουμε προς συζήτηση. Εμείς αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε ήδη από κοινού, δηλαδή ότι η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει, ότι η Ευρώπη έχει μέλλον και οι εθνικοί εγωισμοί δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην αδράνεια. Για τις πιθανότητες ε, εξελίξεων. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό. Αν είχαμε έναν κύριο ευρώ, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Δεν θα έλυνε τα πάντα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν αρκετά χρήσιμο. Για την ομάδα των 20, όταν λέμε ότι οι αγορές θα καθορίσουν τα επιτόκια, τρίχες κατσαρές. Είδαμε τι καθόρισαν οι αγορές μέχρι τώρα. Στην ουσία καταχρηστικές καταστάσεις δημιουργούνται και κάποιοι προσπαθούν να ωφεληθούν από τις ανισότητες τις οποίες οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει απρόβλεπτες εντελώς καταστάσεις. Δεν υπάρχει εν πάση περιπτώσει καμία δυνατότητα πρόβλεψης της αντίδρασης των αγορών έτσι όπως βρισκόμαστε σήμερα. Τώρα για τις αναλύσεις ε, ε, των αιτίων αυτής της ε, κρίσης. Η βασική δυσκολία που έχουμε και είναι μια δυσκολία που παραπέμπει σε συζήτηση με πολιτικούς όρους και εδώ με τον συνόδελφο Έγγελς είχαμε ήδη μια έντονη συζήτηση. Όταν βλέπει κανείς τη στρατηγική του 2020 μπορεί να πει ότι η στρατηγική αυτή δεν προχωρά όσο εμείς θα θέλαμε ή όσο προτείνουμε στην έκθεσή μας αλλά είναι ένα σχέδιο για το τι θα κάνουμε αύριο και έγινε δεκτό από τον Ιούνιο, τον μήνα Ιούνιο επαναλαμβάνω, τον μήνα Οκτώβριο κανονικά το Συμβούλιο θα έλεγε ας βρούμε τρόπους χρηματοδότησης αυτής της στρατηγικής. Τι έκανε, απολύτως τίποτα. Το μόνο που είπε κυρώσεις, κυρώσεις για όλους ουσιαστικά. Το θέμα είναι πώς θα φύγουμε από αυτήν την λογική, πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτά τα μέτρα για το μέλλον. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα πάμε πουθενά. Και αυτή είναι η δύσκολη συζήτηση. Κανένας δεν θέλει να αυξήσουμε τα χρέη, αλλά αν δεν κάνουμε τίποτα κανένας δεν θα μας σώσει από μόνος του. Το να πιστεύει κανείς ότι θα σωθούμε από μια στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουν τα μεγάλα κινέζικα επενδυτικά ταμεία νομίζω ότι αυτό δεν έχει λογική, δεν είναι κάτι το οποίο τεκμηριώνεται. Νομίζω ότι η πρόταση που είχε κάνει η Ντανούτα Χούμπνερ το να υπάρξει μια διάσκεψη δηλαδή λίγο δημόσια αν θέλετε σε σχέση με τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε εμείς είναι μια καλή ιδέα και θα δώσει θα έλεγα σε αυτήν την μακροπρόθεσμη αντίληψη που έχουμε ε, μια κάποια μεγαλύτερη δημόσια ορατότητα και συμφωνούμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Να μην ξεχάσουμε επίσης και ένα συνάδελφος το ανέφερε προηγουμένως ότι πολλά από τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε. Είναι θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε μακροπρόθεσμα και στρατηγικά, από την άλλη όμως είναι θέματα που σε καθημερινή βάση αντιμετωπίζονται από την, κοινωνική, από την οικονομική ε, ε, και νομισματική επιτροπή και εδώ υπάρχει χώρος για κάποιες διευκρινήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώσαμε νομίζω την εξέταση αυτού του θέματος και παρακαλώ τους συντονιστέ να παραμείνουν στην αίθουσα. Ε, τους υπόλοιπους εύχομαι καλή επάνωδο. Καλό βράδυ. Πέντε λεπτά διακοπή και μετά θα αρχίσουμε συνεδρίαση των συντονιστών.